Yeah, it is. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Παρακαλώ καθίστε. Σας καλωσορίζω στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Επιτροπής Απασχόλησης. Προεδρεύω γιατί είμαι, είμαι η μόνη που ε, είμαι στην Επιτροπή από το προηγούμενο Προεδρείο. Πολλοί δεν κατέβηκαν καν σε αυτές τις εκλογές, οπότε δεν επανεξελέγησαν. Ελπίζω να εφαρμόσω σωστά τη διαδικασία. Ε, ελπίζω και εσείς να το χαρείτε. Και ευχαριστώ για την παρουσία σας. Υπάρχει διερμηνία από και προς όλες τις γλώσσες, εκτός από τα Ιρλανδικά, τα γοϊδελικά. Έχουμε και πλήρη και αναπροματικά μέλη. Και κάποιες ανακοινώσεις. Ορισμένων που δεν είναι με αναπροματικά μέλη, αλλά θα ψηφίσουν τώρα S&D, Μάριο Γκρίναου αντικαθιστά τον κύριο, τον κύριο Φούξλαν για το Renew. Η κυρία Βαντράν αντικαθιστά την κυρία Μπόφρη Επίσης, Renew. Η κυρία Ντόνατ αντικαθιστά την κυρία Μάξοβα. Ίσια, Η κυρία Μάζουρε αντικαθιστά την κυρία Νικολασόνοβα. Και από τους μη γεγραμμένους, ο κύριος Λαγός. Αντικαθιστά τον κύριο Νικολάου Αλαβάνο. Νικολάου. Με συγχωρείτε αν δεν τα πρόφερα καλά. Έχουμε 49 συναδέλφους παρόντες, έχουμε λοιπόν απαρτία. Οπότε, άρχεται η συνεδρίαση. Είμαστε εδώ για να εκλέξουμε Προεδρείο για τη νέα θητεία. Το Προεδρείο λοιπόν θα συσταθεί εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τέσσερις αντιπροέδρους και αυτά θα γίνουν με βάση το άρθρο 213 του Συντορικού κανονισμού. Λοιπόν, πρώτα θα λέξουμε τον Πρόεδρο και μετά τους Αντιπρόεδρους. Έχουμε λοιπόν απαρτία, είπαμε. Οπότε, να ρωτήσω εάν υπάρχουν προτάσεις για τον Πρόεδρο, την Προεδρία. Παρακαλώ. Η κυρία Ραβάλσκα. Αγαπητοί συνάδελφοι, από πλευρά του ECA, των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, θέλω να προτείνω την κυρία Βεάτα Σούντλοβ ως πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης απασχόληση και κοινωνικών υποθέσεων. Η κυρία Μπεάτα Σίδλο ήταν πρωθυπουργό της Πολωνίας και πρόεδρο τη Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Εφήρμοσε μια σειρά από κοινωνικές μεταρρυθμίσει στην Πολωνία, οι οποίες μετέβαλαν ουσιοδό την κατάσταση των συμπολιτών μας στην Πολωνία. Ε, αλλαγές στην αγορά εργασίας, της οικογενειακής πολιτικής, και διάφορα άλλα κοινωνικά μέτρα. Οι μεταρρυθμίσει αυτε έκαναν εντύπωση παντού στην Ευρώπη. Κατέδειξαν ότι είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν ε, αποτελεσματικά οι κοινωνικές ανισότητες. Παράλληλα, η κυρία Μπεάτα Σίτλο γνωρίζει, κατανοεί πολύ καλά, το θέμα του κοινωνικού διαλόγου. Συμμετείχε σε κοινωνικό διάλογο με τα συνδικάτα, τις οργανώσεις των εργοδοτών και εκπροσωπώντας πάντα βέβαια την κυβέρνηση. Στον τριμερή αυτό λοιπόν διάλογο. Κατανοεί λοιπόν πολύ καλά την σημασία του διαλόγου και το πόσο σημαντικό να είναι αποτελεσματικός ο διάλογος. Είναι η πεμπτουσία για να επιλύονται τα προβλήματα. Και τα πολιτικά προβλήματα λοιπόν. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τους αδέλφους να στηρίξουν αυτήν την θαυμάσια υποψηφιότητα μιας ε, ιδιαίτερα έμπειρης πολιτικού η οποία ασχολήθηκε με κοινωνικά θέματα ε, για μεγάλο χρονικό διάστημα εστιάζοντας ακριβώς αυτά τα κοινωνικά θέματα. Σας παρακαλώ λοιπόν να την υπερψηφίσετε. Ωραία λέει Πρόεδρος. Οπότε, να ρωτήσω την υποψήφια εάν αποδέχεται την υποψηφιότητα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, την αποδέχομαι και αν μου επιτρέπετε να σας παρουσιάσω το βιογραφικό μου γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί, πολύ να μην με γνωρίζετε αν ε, μου το επιτρέψετε θα ήμουν ε, ευγνώμων. Παρακαλώ λέει ο πρόεδρο, συνεχίστε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη τιμή που προτείνομαι για την Προεδρία αυτή τη επιτροπή. Η Επιτροπή αυτή για μένα είναι από τι πιο σημαντικέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και επειδή ακριβώ έχω πείρα ως ε, Πρωθυπουργό και ε, Αντιπρόεδρος κυβέρνηση έχω ασχοληθεί με πολλά κοινωνικά θέματα. Πολλά θέματα όπου έχουν ε, μεγάλε προσδοκίε οι Ευρωπαίοι συμπολίτε μα Πρέπει να αντιμετωπιστούν λοιπόν και έχουν ήδη γίνει ορισμένα πράγματα. Και σε αυτή την περαιτέρω προσπάθειά μα πρέπει να υπάρχει η αναγκαία βούληση για να δημιουργείται συνένεση. Να υπάρχει ουσιώδης διάλογος. Αυτός είναι ο καλύτερο τρόπο, για να επιτυχάνουμε τι κατάλληλε λύσει για τους συμπολίτε μας ε, που, μες, που μας εμπιστεύτηκαν με αυτή την εντολή να τους εκπροσωπούμε. Σε όλη μου την ε, σταδιοδρομία ασχολήθηκα με κοινωνικά θέματα και ε, της, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης όπου έκανα μια έκκληση για ένα κοινωνικό πρόγραμμα το οποίο εφαρμόσαμε επιτυχώς. Και όπως ανέφερε και η κυρία Ραφάλσκα με την οποία συνεργάστηκα επανειλημμένα. Χάρη και στη δική της βοήθεια εφαρμόσαμε πολλές καλές λύσεις που είχαν ε, θετικό αντίκτυπο και στην Ευρώπη. Ακούστηκαν στην Ευρώπη. Μια έκφραση ε, της αποδοχής ε, της πολιτικής μας από τους συμπολίτε μας ήταν τα αποτελέσματά μας ακριβώς και στις πρόσφατες ευρωεκλογέ. Και η προσωπική μου επιτυχία σε αυτές. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και να εξαλείψουμε τη φτώχεια. Ε, Ιδίω ε, την παιδική φτώχεια και να μειώσουμε την ανεργία η οποία τώρα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επίση, τονίζω ότι χάρη στα προγράμματα αυτά πολλέ κοινωνικέ ομάδε κατάφεραν να βελτιώσουν την κοινωνική του θέση και ζουν τώρα μια καλύτερη ζωή. Είμαι μια περιοχή που υπέφερε κατά τη διάρκεια της ε, οικονομικής μετάβασης και του μετασχηματισμού της οικονομίας αντιμετωπίσαμε πολλές επιπτώσεις στην περιοχή αυτή της συστημικής αλλαγής της πολωνικής οικονομίας. Χάρη σε αυτήν την αλλαγή τώρα η Πολωνία είναι σε πολύ διαφορετική θέση. Εργαζόμενοι λοιπόν σε περιφερειακό επίπεδο κατάλαβα ότι τα κοινωνικά θέματα, τα κοινωνικές ευαισθησίες πρέπει να είναι στην καρδιά της εργασίας ή ουδήποτε πολιτικού. Αν λοιπόν με κλέξετε, αν αποφασίσετε ότι συνεργαζόμενοι μαζί μου ως ε, πρόεδρο, ως πρόεδρο θα με τιμήσετε και σας παρακαλώ να με τιμήσετε με την υποστήριξή σας. Ε, είμαι διατεθειμένη να κάνω διάλογο με όλα τα μέλη της Επιτροπής, με όλες τις πολιτικές ομάδες, γιατί πιστεύω ότι ιδιαίτερα εδώ, σε αυτή την Επιτροπή, πρέπει να είμαστε υπόδειγμα συμπεριφοράς, υπόδειγμα ότι μπορούμε να υπερβαίνουμε τις πολιτικές διαφοροποιήσεις για να εργαστούμε για τα θέματα που αφορούν όλους τους πολίτες και ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ για να εκλεγείτε ως πρόεδρος της Επιτροπής ε, πρέπει να είστε τακτικό μέλος και να έχετε συμπληρώσει την δήλωση οικονομικών συμφερόντων και την δήλωση που αφορά τον ε, κώδικα συμπεριφοράς. Το έχετε κάνει. Οπότε μπορείτε να είστε υποψήφια. Έχω άλλη μία παρατήρηση για τα αναπληρωματικά μέλη. Η κυρία Σάρα Σχίτινταλ αντικαθιστά την Μαρία Βόλς εξ του ΕΛΚ. Οπότε έχουν γίνει όλα αυτά και μπορούμε να περάσουμε στις ε, εκλογές. Κυρία Μπίσοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος ε, της πολιτικής μου ομάδας ε, των Σοσιαλδημοκρατών θα ζητήσω μυστική ψηφοφορία. Μάλιστα. Οπότε, κύριε Κάζα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχουμε ένα σύστημα εδώ, ονόματι DEONT. Και θα έπρεπε να υπάρχει ήδη συμφωνία για τους υποψήφιους και εμείς είμαστε υπέρ αυτού του συστήματος ΔΕΟΝΤ. Αλλιώς θα έχουμε σοβαρές συνέπειες εάν δεν τηρήσουμε την συμφωνία του συστήματος ΔΕΟΝΤ. Όχι μόνο στη δική μας επιτροπή, αλλά και σε άλλες επιτροπές. Οπότε δεν αντιλαμβάνομαι την κίνηση εδώ της σοσιαλίστριας φίλισμου μου όταν έχουμε μόνο μία ε, υποψήφια η οποία αποτελεί άλλωστε αντικείμενο ε, συμφωνίας στο πλαίσιο του συστήματος DEONT για την κατανομή των αξιώματων. Δεν βλέπω τον λόγο να έχουμε μυστική ψηφοφορία, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε και πρέπει να δείξουμε στο ευρωπαϊκό κοινό ότι έχουμε ένα σύστημα εδώ το οποίο ε, τηρούμε και τηρούμε τις συμφωνίες που προκύπτουν από αυτό. Οπότε μυστική ψηφοφορία για κάτι το ήδη συμφωνημένο δεν ξέρω αν είναι το σωστό μήνυμα προς τα έξω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πιτζλάρο ζητάει λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, πράγματι θεωρώ ότι ο κύριος Ντεόντι ήταν ε, ιδιοφυΐα, μαθηματικός και βεβαίω ε, δεν βρισκόμαστε εδώ πέρα χάρη μαθηματικών υπολογισμών, αλλά χάρη των υπολογισμών των ψήφων. Και έχουμε νομίζω την νομοποίηση να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Δεν είναι θέμα του να μην επιτρέψουμε κάποιον υποψήφιο, είναι θέμα του να επιλέξουμε μία διαδικασία. Δεν είναι ζήτημα του να κρύψουμε κάτι. Εγώ στηρίζω λοιπόν την πρόταση των σοσιαλδημοκρατών για μυστική ψηφοφορία. ευχαριστώ. Ε, απαιτούνται 11 βουλευτές για μυστική ψηφοφορία. Έχουμε πάνω από 11, οπότε πάμε σε μυστική ψηφοφορία για αυτήν την υποψηφιότητα και εδώ πρέπει να πω ότι για την ψηφοφορία αυτήν μπορείτε βεβαίως ε, πάντα να επιλέξετε την αποχή, αλλά δεν μετράει. Θα μετρήσουμε τα υπέρ και τα κατά. Το πράσινο κουμπάκι είναι υπέρ, το κόκκινο κουμπί είναι κατά άρχια η okay, there are, there are, there are three too many EPP. Τρεις παραπάνω ψηφίζουν από το ΕΛΚ. Ψηφίζουμε ε, την υποψηφιότητα. Αν είστε υπέρ της υποψηφίου πατάτε το πράσινο, κατά πατάτε το κόκκινο. Και τώρα, εντάξει. Ωραία, ευχαριστούμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Ως αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έχουμε 21 υπέρ, 27 κατά, δύο αποχές. Οι αποχές δεν μετράνε, αλλά η υποψήφια δεν εκλέγεται, οπότε προτείνω να ε, Διακοπή εδώ η συνεδρίαση και να επαναληφθεί κάποια άλλη στιγμή. Συμφωνείτε κύριε Κάζα ε, να αναβληθεί εννοείται μέχρι την επόμενη εβδομάδα για να βρεθεί χρόνος για να βρούμε μία λύση σε αυτό το μοναδικό πρόβλημα. Η πρότασή μου είναι να διακοπεί η συνεδρίαση και να ζητήσουμε από τη γραμματεία να μας βρει ε, μια άλλη χρονική στιγμή. Συμφωνείτε? Ωραία. Λοιπόν, λίγα τη συνεδρία. Ευχαριστώ.